Uh, Καλημέρα σε όλους. Κυρία Υπουργέ, με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζω στην συνεδρίαση της υποεπιτροπής μας και να ευχαριστήσω και τον κύριο Νταντζάν που είναι πρόεδρος της υποεπιτροπής που οργάνωσε αυτή τη συνάντηση μαζί σας. Ξέρετε ότι η επίσκεψή σας είναι ιδιαίτερα επίκαιρη όχι μόνο λόγω τη ουσία του θέματο των προτεραιοτήτων της Ισπανική Προεδρία, αλλά όπω ξέρετε αρχίζουμε να ασχολούμαστε και με τι συνέπειε τη υλοποίηση τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Προφανώ λοιπόν θα καταβληθούν ιδιαίτερε προσπάθειε για να εξέφερουμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ των όσων επιτάσσει η συνθήκη και της πραγματικότητας εντός της οποίας θα πρέπει να την εφαρμόσουμε. Με ναι, αυτά τα λόγια θα ήθελα να ζητήσω από τον κύριο Νταντζάν τον πρόεδρο της Υποεπιτροπής, να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε σε αυτή την ε, παραδοσιακή συνάντηση της ασκούσας προεδρίας με την ε, υποεπιτροπή μας. Όπως θύμισε ο συνάδελφος Πασκού, είναι μια σημαντική στιγμή διότι τώρα ζούμε την πρώτη, τις πρώτες φάσεις της εφαρμογής της συνθήκης της Λισαβόνας που έχει συνέπειες για την πολιτική ασφαλείας και άμυνας, αλλά και από συγκυριακής άποψης είναι κατάλληλη στιγμή, γιατί υποδεχτήκατε την πάλμα του 27 υπουργού άμυνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπήρχε και μια σοβαρή απουσία τις ημέρες εκείνες Και σήμερα είναι σημαντικό να έχουμε την παρουσία σα εδώ, καθώς και τα... το λόγο σα στην δική σα την άποψη μετά τη σιωπή των τελευταίων ημερών και των τελευταίων εβδομάδων. Μια δική μα αντιπροσωπεία μετέβη στη Μαδρίτη στα τέλη Δεκεμβρίου και είχε μια ιδιαίτερα επικοδομητική και καρποφόρα συζήτηση με του εκπροσώπου του Υπουργείου σα για τι προτεραιότητε τη δική σα Προεδρία στα θέματα ασφάλεια και άμυνα. Με ιδιαίτερη χαρά λοιπόν σα ακούμε σήμερα και σα δίνω το λόγο για να μα κάνετε την παρουσίαση σα. Ευχαριστώ. Καλημέρα, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι μεγάλη μου ευχαρίστηση αλλά και τιμή να έρχομαι εγώ για να σας ε, μιλήσω και να σας πω ποιες είναι οι προτεραιότητες πλευράς ασφάλειας και άμυνας της Προεδρίας της Ισπανίας. Είναι μεγάλη μου τιμή, επαναλαμβάνω, που με προσκαλέσατε σήμερα εδώ. Όπω ξέρετε, για τέταρτη φορά αναλαμβάνουμε την ε, κυκλικά αναλογούμενη την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το, 1986, 86 όταν μπήκαμε στην τότε ΕΟΚ ε, δείξαμε ότι είμαστε αποφασισμένοι ε, για μια Ευρώπη ολοκλήρωσης, καινοτομίας, ανταγωνισμού, αλληλεγγύης για την Ευρώπη των πολιτών, αλλά και ασφάλειας και άμυνας ανέκαθεν θέλαμε να βοηθήσουμε για να είμαστε πρωτοπόροι όσον αφορά μια πολιτική άμυνας και ε, όσα χρόνια υπάρχει ε, κάναμε ό,τι μπορούσαμε ε, στα πιο καυτά σημεία του πλανήτη. Έχουμε 23 αποστολές μέχρι τώρα και γι' αυτό το λόγο έχουμε και την πείρα που χρειάζεται αλλά επίσης έχουμε και τις δυνατότητες ούτως ώστε να αντιμετωπίσουμε τις νέες προκλήσεις αλλά και απειλές. Όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος Αντιπρόεδρος, ε, σε πάρα πολύ κρίσιμη στιγμή και συγκέντρωση οικοδόμησης να λαμβάνουμε αυτή την ε, Προεδρία όσον αφορά και την ε, Συνθήκη της Λισαβόνας που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση η Ευρωπαϊκή Ένωση και ως μια δύναμη κοινωνική, οικονομική αλλά και σαν έναν πρωταγωνιστή στη διεθνή σκηνή όσον αφορά τη διατήρηση της ειρήνης και επίσης Έχουμε τώρα κάποιες καινοτομίες από πλευράς ασφάλειας που ήδη γνωρίζετε, οπότε δεν χρειάζεται να επιστρέψω σε αυτές τις λεπτομέρειες. Έχουμε την καινούργια ΚΕΠΑ που θα είναι κάτι πάρα πολύ βασικό, ώστε να μπορέσουμε τα όσα έχουμε μέχρι τώρα πετύχει να τα ε, στεριώσουμε, να τα παγιώσουμε και να μπορέσουμε να δράσουμε και στη διεθνή σκηνή και στο εσωτερικό της Ένωσης. Αυτή η κοινή πολιτική είναι ένα βήμα προς τα εμπρός, για να ολοκληρωθεί και η Ευρώπη της Άμυνας. Έχουμε επίσης αυτές τις ρήτρε της ελληνικής και της αμοιβαία αρρωγής. Επίσης υπάρχει δυνατότητα να έχουμε μία διαρθρωμένη μόνιμη συνεργασία και συνεργασία ενισχυμένη, ούτως ώστε να μπορέσουμε να διαχειριζόμαστε τις κρίσεις ε, και να έχουμε στα χέρια μας τα εργαλεία που χρειάζονται για αυτό το λόγο. Επίσης, σύμφωνα με την συνθήκη, έχουμε κάποιες συγκεκριμένες διατάξεις όσον αφορά μία την υπηρεσία άμυνας, ε, ιδίω έχουμε το θέμα για την εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών, ε, να προωθηθεί η έρευνα, ε, τεχνολογική βάση, η βιομηχανία να βοηθήσει επίσης και επίσης όσον αφορά τις στρατιωτικές δαπάνες αλλά και την άριστη αξιοποίηση των πόρων. Μπορούμε με τη συνθήκη να έχουμε νομική βάση, μπορούμε να έχουμε ξεκάθαρα μέσα πολιτικής και πολύ συγκεκριμένα, ούτω ώστε να μπορέσουμε αυτήν την ΚΕΠΑ να την εξελίξουμε και να την προωθήσουμε. Επίσης έχουμε τον, ε, τη συνεννόηση με, με την υψηλή εκπρόσωπο και στη συνέχεια ε, ε, να σας πω πιο συγκεκριμένα πράγματα της πολιτικής μας έχουμε ως κριτήρια της πολιτικής μας την συνένεση, τον ρεαλισμό αλλά και την ευελιξία. Και με αυτά τα κριτήρια θα έχουμε έναν μπούσουλα ούτω ώστε στην πολιτική μας να μπορέσουμε να βάλουμε ένα λιθαράκι παραπάνω, να είναι μια προσθεμένη αξία όλα αυτά τα οποία κάνουμε και έτσι να μπορέσουμε να κάνουμε κάποια βήματα προς τα εμπρός συγκεκριμένα και βιώσιμα. Ε, με τη συνεργασία επομένως και τη βοήθεια από την υψηλή εκπρόσωπο θα, έχουμε τα εξής. Θα κινηθούμε στα θεσμικά ζητήματα, ανάπτυξη των δυνατοτήτων της Ένωσης, αλλά και ε, μια ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των κρίσεων. Στην τελευταία συνάντηση την άτυπη των Υπουργών στην ε, Πάλμα, στη Μαγιόρκα, 24 και 25 Δευτέρου, επιβεβαιώθηκαν αυτές οι προτεραιότητες που θα σας ε, αναπτύξω. Ο πρώτος άξονας θεσμικά ζητήματα. Η συνθήκη, όπως γνωρίζετε, τώρα δίνει περισσότερες αρμοδιότητες στους υπουργούς άμυνας και ευξημένες αρμοδιότητες λήψης αποφάσεων. Γι' αυτό και εμείς έχουμε ως στόχο να μπορούμε να ενισχύσουμε αυτές τις, ε, τις, ε, τις συναντήσεις των Υπουργών επί τη βάση της συνθήκης. Επίσης, στην ε, Μαγιόργα οι Υπουργοί Άμυνας συμφώνησαν ότι θα πρέπει στι συναντήσει να λαμβάνονται αποφάσει όσον αφορά την ανάπτυξη των δυνατοτήτων τη Ένωση, όσον αφορά τι ε, ευρωπαϊκέ δυνάμει, το προσωπικό, του πόρου που χρειάζονται για την Ευρώπη τη Άμυνα, Επίση, συμφωνήσαμε όσον αφορά την αμοιβή αρρωγή αλλά και την ρήτρα ελληνική, Για να μπορούμε όλα αυτά να τα υλοποιήσουμε, απευθυνθήκαμε στην υψηλή εκπρόσωπο θα πρέπει η υψηλή εκπρόσωπος, η να κατεβάσει συγκεκριμένε προτάσεις στο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών. Τον Απρίλιο θα γίνει μια τέτοια συνάντηση στο Λουξεμβούργο. Επίσης, όσον αφορά τις δυνατότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είμαι θα πεπισμένη ότι είναι δυνατόν και πρέπει να επιφέρουμε κάποιες βελτιώσεις. τελειώνει το πρόγραμμα για, την πολιτική μας που υπήρχε το 2010, επομένως θα πρέπει να κάτσουμε κάνουμε έναν απολογισμό του τι πετύχαμε και επίσης να προβληματιστούμε για το μέλλον και να δούμε πώς θα άρουμε τις αδυναμίες που έχουν παρατηρηθεί. Και βεβαίως θα πρέπει να δούμε πώς θα γίνουμε πιο αποδοτικοί. Όσον αφορά τώρα το τι μπορεί να κάνουμε όσον αφορά την άμεση και ταχεία αντίδραση ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεωρεί η Προεδρία ότι υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία είναι δυνατόν και πρέπει να βελτιωθούν. Και έτσι να είναι δυνατόν να χρησιμοποιούμε καλύτερα αυτή τη δυνατότητα της ταχείας επέμβασης. Θα γίνει ένα σεμινάριο εδώ για να δούμε πώς μπορούμε να έχουμε κάποιο είδους επανεμβάσεις ε, αυτές τις, τις ομάδες ταχείας ε, ανάπτυξης, πώς μπορεί να γίνεται πιο γρήγορα, πώς μπορεί να γίνει η χρηματοδότηση. Και επίσης θα πρέπει να σας πω ότι στην Μαγιόρκα την περσμένη εβδομάδα ενέκριναν οι Υπουργοί Άμυνας αυτήν την βελτίωση της δυνατότητας αυτών των, των ταχαίων δυνάμεων επέμβασης, ούτως ώστε να μπορούμε να διαχειριστούμε κάποιε. Ε, ανθρωπιστικές ε, ε, κρίσεις, να διαχειριστούμε κάποιες θεομηνίες και να έχουμε μόνο σε αυτό το εργαλείο και σαν Ευρώπη να μπορούμε άμεσα να κάνουμε κάτι όταν υπάρχει κάποια ανθρωπιστική κρίση, κάτι το κατεπήγον, κάποια καταστροφή. Οπότε γι' αυτό και θεωρούμε ότι ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Αμήνα θα πρέπει να δει πώ μπορεί επί τη βάση τη Συνθήκη Λισαβόνα να αναπτύσσει δραστηριότητέ τη και μόλι ολοκληρωθεί αυτό ο, ο στόχο του 2010, εκείνο το πρόγραμμα, θα δούμε πώ θα βελτιώσουμε την άμυνα, πώ θα βελτιώσουμε τον εξοπλισμό, πώ θα βελτιώσουμε τη διαχείριση κάποιων προγραμμάτων επί τη βάση τη ε, βιομηχανία άμυνα τη Ευρώπη. Και γι' αυτό έχουμε οργανώσει δύο σεμινάρια πρώτα-πρώτα. Ε, Συνέργειε για ανάπτυξη των πολιτικών αλλά και στρατιωτικών τρόπων διαχείρισης κρίσεων στην Ευρώπη. Αυτό στη... έγινε στις Βρυξέλλες και επίσης και για ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ πολιτικών αρχών και στρατιωτικών αρχών. Το πώς είναι δυνατόν να είναι δυνατόν να συγκλίνουν ε, οι σχετικές υπηρεσίες για, ε, για τέτοιου είδους ε, αντιμετώπιση κρίσεων. 16 Φεβρουαρίου στη Μαδρίτη Επίση, διαχείριση προγραμμάτων είχαμε και διαχείριση του εξοπλισμού. Ένα άλλο σεμινάριο. Θα γίνει τώρα το Μάρτιο ένα άλλο σεμινάριο όσον αφορά την αναδιάρθρωση τη ε, βιομηχανία άμυνα. Και θα δούμε τι, τι μπορούμε να έχουμε όσον αφορά την καινοτομία και έτσι να δούμε πώ θα μπορέσουμε να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί σε αυτό τον τομέα. Επίση, όπω προείπα, ε, θα πρέπει να δούμε πώ θα έχουμε μια διαρθρωμένη, μόνιμη δομημένη συνεργασία. Και έτσι θα πρέπει να ξεκινήσουμε τις αρχικές συνομιλίες. Γι' αυτό και θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξεκαθαριστεί το ποιοι είναι οι στόχοι αυτής της ε, συνεργασίας και ιδίως να δούμε με ποιους μηχανισμούς μπορούμε όλα αυτά να τα υλοποιήσουμε στις 16 Τρίτου. Εδώ στις Βρυξέλλες θα οργανώσουμε ένα σεμινάριο για να μπορέσουμε να συζητήσουμε το θέμα τούτο. Βεβαίως και πρόκειται τα συμπεράσματα να διαβιβαστούν στην ύπατη εκπρόσωπο, ούτω ώστε να ληφθούν όλα αυτά υπόψη. Τέλος, τι γίνεται με το στρατιωτικό μας προσωπικό, άνδρες και γυναίκες που υπηρετούν στις στρατιωτικές μας ε, δυνάμεις και που υλοποιούν την ΚΕΠΑ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούν αυτοί να ξέρουν τι γίνεται, να ξέρουν και τα θεσμικά και τα νομικά ζητήματα που υπάρχουν. Και για να διευκολύνουμε κατά την κατάρτιση των ε, αξιωματικών του προσωπικού κάνουμε στις σχολές ευελπίδων, στις στρατιωτικές μας σχολές, σεμινάρια για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις και για την ΚΕΠΑ πιο συγκεκριμένα και το ίδιο ε, ίσως θα πρέπει να γίνεται και σε όλα τα κρατημέλη θα μπορέσουμε με αυτόν τον τρόπο να βελτιώσουμε τις δυνατότητες ε, και αυτών των ομάδων ταχείας επέμβασης και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Άμυνας. Είναι κάτι το οποίο βρήκε σύμφωνος όλους τους υπουργούς στη συνάντηση που έγινε στην Πάλμα, στη Μαγιόρκα. Πέραν των θεσμικών ζητημάτων, πέραν ε, των δυνατήτων της Ένωσης και της αναβαθμισής τους, εμείς Θέλουμε να έχουμε μια ολοκληρωμένη οπτική της πολιτικής της ασφάλειας, άρα χρειάζεται συντονισμός, χρειάζεται συνεργασία και με τους άλλους ε, εμπλεκομένους στα διάφορα επίπεδα όπου λειτουργεί η πολιτική μας και γνωρίζουμε ότι η διαχείριση και η αντιμετώπιση των κρίσεων προαπαιτεί συνδυασμό στρατιωτικών και πολιτικών δυναμιών. Και η Σουηδική Προεδρία κατάφερε μια τέτοια συνέργεια για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων μας. Και εμείς θα κάνουμε το ίδιο και θα προσπαθήσουμε να προωθήσουμε ακόμα περισσότερο ε, αυτές τις δυνατότητες. Και για την ασφάλεια των θαλασσών θέλουμε συνεργασία μεταξύ πολιτικών θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, η ΚΕΠΑ είναι θέμα του Συμβουλίου, αλλά θα πράττουμε και τι θα γίνει όσον αφορά την γενικότερη πολιτική για τις θάλασσες, που είναι θέμα και αρμοδιότητα της Κομισιόν. Τώρα το, αυτό το Μάρτιο θα κάνουμε ένα ακόμα σεμινάριο στη Μαδρίτη όσον αφορά την ασφάλεια στις θάλασσες για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να δούμε ποια είναι τα βασικά στοιχεία ούτως ώστε να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ασφάλεια στις θάλασσες. Καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών χρειάζεται. Επίσης να υπάρχει μια αμοιβαία εμπιστοσύνη, ε, αναβάθμιση των δυνατοτήτων όλων των εμπλεκομένων και προσαρμογή αυτών στις νομικές βάσεις που έχουμε. Συμφωνήσαμε οι Υπουργοί στη Μαγιόρκα να υπάρχει μια ομάδα εμπειρογνωμόνων Συμβουλίου και Κομισιών. Από κοινού αυτοί οι εμπειρογνώμονες να δουν πώς θα έχουμε ασφάλειες θάλασσες και μια σχετική πολιτική που να συνδυάζει στρατιωτικά και πολιτικά μέσα και στο Λουξεμβούργο θα συγκροτηθεί σχετική ομάδα εργασία. Στα πλαίσια αυτή τη ασφαλεία για τη θάλασσα θέλουμε να αντιμετωπίσουμε βεβαίω και την πειρατεία. Ε, και αυτό να γίνει σε κλίμακα παγκόσμια. Έχουμε βέβαια την επιχείρηση Αταλάντη όσον αφορά τις ακτές της Σομαλίας. Επίσης, Το Μάιο θα έχουμε ένα συμπόσιο, μια εκδήλωση για το ίδιο θέμα, όπου θα προσκληθούν πάρα πολλοί διεθνεί φορεί. Θεωρούμε ότι είναι προτεραιότητα τη Προεδρία μα να έχουμε καλύτερη συνεργασία και συντονισμό και με του άλλου εμπλεκομένου στο θέατρο των επιχειρήσεων, για αυτό το λόγο. Οπότε και εξετάζουμε ποιε είναι οι αλλακτικέ για, για να υπάρχει τεχνική συνεργασία με το ΝΑΤΟ. Στη Μαγιόρκα αποφάσισαν οι υπουργοί το θέμα αυτό να το συζητήσουμε με τον ε, κύριο Ράσμουσεν, τον ε, ΓΓ του ΝΑΤΟ, οπότε συμφωνήσαμε ότι χρειάζεται να υπάρχει ένα πλαίσιο μόνιμης πάγιας συνεργασίας μεταξύ ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης, όποτε υπάρχει λόγος ε, κοινού θεάτρου επιχειρήσεων για να μπορούμε να εκμεταλλευτούμε καλύτερα και να συνδυάσουμε τις δυνατότητες ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε χρειάζεται καλύτερη συνεργασία. Ε, να αναβαθμίσουμε τις δυνατότητες τις μεταφορικές και να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις αυτοσχέδιες βόμβες που είναι η μεγαλύτερη απειλή για το προσωπικό μας. 16 Τετάρτου στην ε, Μαδρίτη επίσης θα γίνει μια εκδήλωση για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να έχουμε πιο πάγιες δομές συνεργασίας για διαχείριση κρίσεων μεταξύ Ένωσης και ΝΑΤΟ και επομένως να έχουμε εναρμονισμένη λειτουργία ε, των μηχανισμών των δυνατοτήτων μας. Επίσης, τον Ιούνιο θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ε, μια, μια εκδήλωση, ούτω ώστε να δούμε πώς μπορεί να γίνει χρήση ελικοπτέρων σε παιδινά, ορεινά, μειωρινά εδάφη για όποτε χρειάζεται. Όπως είπαμε και για τις βόμβες, θα δούμε πώς μπορεί να γίνεται η απενεργοποίησή τους ε, από πλευράς πυροτεχνουργών και στο Μανθανάρα θα υπάρχει εκεί πέρα μια συνάντηση ούτω ώστε να δούμε πώς θα συνδυαστεί και σε αυτή την περίπτωση ε, η πώς θα συντηρηθούν οι δυνατότητε Ένωση και ΝΑΤΟ. Επίσης και με τρίτες χώρες να υπάρχει συνεννόηση, επομένως ε, στο, στο, στο περιθώριο της συνάντηση της Μαγιόρκα ε, συναντήσαμε εκπροσώπου των χωρών ε, της Νοτίου ε, Μεσογείου, Τίνιδα, Μαρόκο, Μαυρετανία, ε, Αλγερία, Λιβύη, οπότε έτσι προσπαθήσαμε να δούμε πώς βλέπει ο καθένας τις απειλές ε, του, του κοινό εχθρό και να δούμε πώς σε τακτική βάση θα συναντιόμαστε για να αναζητούμε λύσεις αντιμετώπισης. Επίσης, θα δούμε πώς θα συνεχίσουμε τις αποστολές που τώρα βρίσκονται την εξέλιξη και ε, πώς θα γίνει ο συνδυασμός ε, πολιτικών και στρατιωτικών γι' αυτό. Αλτέα, στην Βοσνία Ριζεγοβίνη Συμφωνούμε όλοι ότι ήταν πετυχημένη επιχείρηση και ότι υλοποιήθηκαν οι στόχοι της συμφωνίας του Ντέιτον. Σήμερα η λειτουργία εκεί είναι κυρίως πολιτική. Ο καλύτερος τρόπος για να βοηθήσουμε σήμερα την Βοσνία Ζεγοβίνη είναι να στεριώσει εκεί η ειρήνη και να πλησιάσει και γιατί όχι μια μέρα να ενταχθεί σε ΟΚ και ΝΑΤΟ. Επομένω θα πρέπει να προχωρήσουν οι αναγκαίε μεταρρυθμίσει. Στη Μαγιόρκα, οι Υπουργοί Άμυνα μελέτησαν τι αποφάσει 25 Ιανουαρίου των Υπουργών Εξωτερικών όσον αφορά μια αποστολή που θα αξιολογήσει στην Βοσνία Ζεγοβίνη πώ έχει η κατάσταση από και στρατηγική πλευρά. Τα κράτη-μέλη είπαν ότι επιθυμούν να συνεχιστούν οι συνομιλίε για το μέλλον της Αλτέα. Αυτό θα γίνει τον Απρίλιο στο Συμβούλιο του Λουξεμβούργου και κατόπιν ε, θα γίνει μια αποστολή το φθινόπωρο επιτόπου. Αταλάντη. Ακτές Σομαλίας. Εκεί έχουμε λένε και περισσότερα επεισόδια πειρατείας και λένε και περισσότερα ανησυχεί διεθνείς κοινότητες η επιχείρησή μας μείωσε τις πειρατικές επιθέσεις και τις απαγωγές. Ε, Ήταν μία στις τρεις επιθέσεις που κατέληγαν σε απαγωγή, τώρα είναι μία στις έξι. Έχουμε μόνο σε αυτά τα κομβόη, τα οποία τώρα προστατεύονται, τα κομβόη της ανθρωπιστικής βοήθειας. Και γενικότερα προσπαθούμε να προστατεύσουν εμπορικά πλοία στον ε, κόλπο του Άντεν. Όμως, αυτό επιδέχεται βελτίωση. Άρα θα πρέπει να πάρουμε κάποια μέτρα για να βελτιώσουμε την επιχείρηση και για να μπορέσουμε να, να επαναπροσανατολίσουμε την επιχείρηση Αταλάντη σύμφωνα με την κτηθήσα εμπειρία. Κατά την συνάντηση της Μαγιόρκα, οι Υπουργοί συμφωνήσαμε στο ότι θα πρέπει να δούμε ποιε είναι οι επιλογέ σύμφωνα με του επικεφαλεί τη επιχείρηση, να επαγρυπνούμε, να ελέγχουμε τα ε, λιμάνια τις βάσεις των πειρατών, να τις ε, ψάχνουμε ε, και να δούμε πώς θα εξουδετερώνουμε τα πειρατικά πλοία. Και να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε τις πράξεις πειρατείας ακόμα και χίλια μίλια από την ακτή. Γιατί αυτό κάνουν οι πειρατές. Έχουμε με την Κένια κάποιες ε, συμφωνίες και θα πρέπει να κάνουμε και με την ε, Τανζανία, τον, τον Μαυρίκιο, την Νοτιοαφρικανική Δημοκρατία, τις σχετικές ε, συμφωνίες, ώστε να πλησιωθεί η δράση μας με αυτές τις συμφωνίες. Όλοι στην Μαγιόρκα επίσης συμφωνήσαμε ότι θα πρέπει στο Λουξεμβούργο να συζητηθεί και να ληφθεί επίσημη απόφαση όσον αφορά την παράταση της λειτουργίας της επιχείρησης Αταλάντη για το επόμενο έτος. Όλοι συμφωνούμε. Και για να, αν θέλουμε να είμαστε θα πρέπει να υπάρχει μια επαόριστον ε, παράταση. Και πολλές φορές χρειάζεται συνδυασμός δράσης και στην ξηρά. Υπάρχει πρόβλημα με τη Σομαλία όσον αφορά τι απαγωγέ των πλοίων και γι' αυτό συμφωνήσαμε να συνεχιστεί μια διαδικασία, η διαδικασία που προβλέπεται για την, για την ασφάλεια στη, στη Σομαλία και για ακόμα μία χρονιά και ότι έτσι να έχουμε περισσότερες δυνατότητες επιχειρησιακές και αυτό θα επισφραγιστεί σαν απόφαση τον Μάιο. Πρωτοπόροι ήμασταν επίσης όσον αφορά ε, την αναγνωριστική δράση εκεί, μια ομάδα επιχειρησιακή επιτελική εδώ στις Βρυξέλλες και επίσης ε, θα στελεχώσουμε και τους επικεφαλείς των, των επιτελείων επιτόπου και στις Βρυξέλλες, στις σχετικές υπηρεσίες. Επομένως, θα συνεχιστεί η λειτουργία ε, αυτή η επιχειρησιακή που ξεκίνησε τον Νοέμβριο. Τέλος, θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε όσον αφορά αυτή την θεομηνία που έπληξε την, ε, την IT. Σε συνδυασμό με διάφορους φορείς και την κυβέρνηση της χώρας, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέπτυξε και εκεί ε, ό,τι, ό,τι τη ζητήθηκε από τα μέσων, ανθρωπίνων πόρων κλπ. Ούτω ώστε να προστατευθεί ο κόσμος, να φτάσει και ανθρωπιστική βοήθεια, ε, ε, να υπάρχει και κάποια προσπάθεια για ασφάλεια. Οπότε, με πρόταση τη εκπροσώπου, όπω γνωρίζετε, εδώ στι Βρυξέλλε, οι υπουργοί συγκρότησαν μια ομάδα συντονισμού για την ΑΕΤ. Οπότε έχει ένα κέντρο εκεί ελέγχου και ενημέρωση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμεί ε, είμαστε ελέγχοι ε, βέβαια, με τον ΑΕΤΙΝΟ λαό και ω Προεδρία βοηθήσαμε, προωθήσαμε διάφορε πρωτοβουλίε, τόσο ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε για την αντιμετώπιση αυτή τη τρομερή κατάσταση και επομένω η δράση τη Ένωση ήταν ένα πράγμα προ μίμηση. Πώ μπορούν τα κράτη-μέλη όταν θέλουν, όταν συντονιστούν να πετύχουν πολλά. Επομένω ήταν πάρα πολύ καλά όλα αυτά ε, και αλλά θα πρέπει φυσικά να δούμε πώ μπορούμε να είμαστε ακόμα πιο αποδοτικοί, ακόμα καλύτεροι. Στη Μαγιόρκα Επίσης προτείναμε να βελτιωθεί η άμεση επέμβαση σε κρίσεις και ανθρωπιστικές κρίσεις. Όλοι οι υπουργοί συμφώνησαν ζητήσαμε από την υψηλή εκπρόσωπο να κατεβάσει κάποιες προτάσεις και αυτές να συζητηθούν τον Απρίλιο στο Λουξεμβούργο. Νομίζω πρέπει να συμπεράσματα από την εμπειρία μας και κυρίως από την ε, IT. και να δούμε αν έχουμε τα κατάλληλα εργαλεία πολιτικής στη διάθεσή μας, μέσα πολιτικής, τόσο ώστε να μπορούμε να παρέμβουμε σε καταστροφές και σε κρίσεις όπως θέλουμε, όσο άμεσα θέλουμε. Είναι κατακλείδη. Γι' αυτό το εξάμεινο η Προεδρία θέλει να ενδυναμώσει, να αναβαθμίσει το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διεθνή σκηνή, ούτω ώστε να μπορούμε να παρουσιάσουμε αντίστοιχη του οικονομικού μας μεγέθους. Από πλευρά ασφάλειας και άμυνας πάμε προς την επίτευξη αυτού του στόχου. Έχουμε τα, μέσα, τα, τα θεσμικά, έχουμε κάποιους στόχους, οπότε θα πρέπει να έχουμε ένα πρόγραμμα εργασίας για τους ε, στόχους που έχουμε, για τις προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και γι' αυτό και κάναμε και αυτά τα σεμινάρια που σας είπα ε, και αντίστοιχα τα συζητήσαμε αυτά στην ε, Μαγιόρκα και συμφωνήθηκε κάθε μία από αυτές τις προτάσεις που κατεβάσαμε. Πάρα πολύ χρήσιμα ήταν και τα σεμινάρια για την Προεδρία πάντως, γιατί μπορέσαμε να έχουμε προσέγγιση στις επιμέρους θέσεις, να διευκολυνθεί η λήψη αποφάσεων για τα διάφορα ζητήματα. Θα συνεχίσουμε να προαγάγουμε τις πρωτοβουλίες που, που, έχουμε για να κορυφωθεί αυτή η διαδικασία στο Λουξεμβούργο, γιατί είναι όλα αυτά πάρα πολύ σημαντικά ε, ασφάλεια στη θάλασσα, αναβάθμιση δυνατοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, όλα αυτά θέλουμε ότι είναι υποχρέωσή μας και όπως ε, ανέφερα στην αρχή. Θέλουμε και δεσμευόμαστε να προωθήσουμε μια πιο ολοκληρωμένη ΚΕΠΑ και να μπορούμε να μπορούμε οι αξίες μας για την ε, αλληλεγγύη και, και, οι υπόλοιπε να μεταλαμπαδεύονται σε όλο τον κόσμο. Σούμαν, Μονέ και οι άλλοι πατέρε τη Ευρώπη θέλανε να είναι ε, η Ευρώπη ολοκληρωμένη παντού, οικονομικά, πολιτικά και πλευρά άμυνα. Ευρώπη σημαίνει ειρήνη. Αυτό σημαίνει ευρωπαϊκή οικοδόμηση, είπε ο Ζόμονε. Και επομένω για άμυνα και και ασφάλεια. Θέλουμε να προωθήσουμε την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Δεσμευόμαστε και εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Θεωρούμε ότι είναι ευθύνη και υπευθυνότητά μας. Ευχαριστούμε κυρία Υπουργέ για αυτό το πολύ κατατοπιστικό πανόραμα, την πανοραμική εικόνα των πρωτοβουλειών που μας παρουσιάσατε. Χαιρετίζω ιδιαίτερος το έργο που θέλετε να φέρετε εις πέρας για την μόνιμη διορθωμένη δομή. Μια τη τις που προβλέπει η συνθήκη, αλλά που παραμένει για την ώρα αφηρημένη έννοια. Εδώ στο Κοινοβούλιο ακριβώς καλούμεθα να συζητήσουμε ενδελεχώς και να μελετήσουμε αυτό το θέμα. Επίσης και για το θεσμικό πλαίσιο, για τις δυνατότητές μας, για το επιχειρησιακό σκέλος. Μας μιλήσατε διαμακρών. Έχω και εγώ, όπως και πολλοί συνάδελφοι, κάποιες ερωτήσεις. Μία πρώτα απ' όλα θεσμικού χαρακτήρα. Είπατε ότι πρέπει να ενισχυθούν οι συναντήσεις των κεφαλής άμυνας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό συζητήθηκε και στην Πάλιμα της Μαγιόρκα. Εσείς πώς ελπίζετε στο μέλλον να οργανωθεί αυτό. Θα υπάρξει ένα αυτό καθεαυτό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Υπουργών Άμυνα, στο οποίο θα προεδρεύει η κυρία Άστον. Είναι μια ιδέα την οποία διαβλέπετε να ελοπείτε στο μέλλον και έπειτα για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνα. Αναπτύξατε ένα θέμα που για μας είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον για τους δυνατότητε που θα έχει ο οργανισμός αυτό και για το ρόλο του οργανισμού που έχει αναγνωριστεί και με τη νέα συνθήκη. Ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν υπάρχει όμω ομοφωνία για το ρόλο που θα πρέπει να αναλάβει αυτός ο οργανισμός μεταξύ των κρατών μελών και για τα μέσα με τα οποία θα προοικοδοτηθεί ο οργανισμό. Να κάτι που πρέπει να μελετήσουμε επίση και κάτι που είχε τεθεί και στην ύπατη εκπρόσωπο εδώ και είχε εκφράσει και μια σχετική επιφυλακτικότητα για το όλο θέμα. Εσείς πώς θα το βλέπατε το ζήτημα αυτό. Είναι οι δικές μου δύο ερωτήσεις αυτές. Και τώρα να δώσω το λόγο στον Αντιπρόεδρο, τον κύριο Πασκού, ο οποίος θέλει και εκείνος να παρέμβει. Thank you very much and... Σας uh, <coughs> ευχαριστώ. Να σας ευχαριστήσω και εγώ για την παρουσίαση αυτή, που ήταν πραγματικά εκτενής και μας ε, δίνει μία ένδειξη για τις προθέσεις σας, ιδιαίτερα στη στιγμή αυτή, όπου καλούμαστε να εφαρμόσουμε τη συνθήκη της Λισαβόνας. Θα γνωρίζετε ότι νομίζω ότι εξετάζουμε ιδιαίτερα τα, τη μηχανική των καταστάσεων, πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τη μηχανική, αλλά ξέρετε πολλές φορές χάνουμε την πολιτική διάσταση Και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να κοιτάξουμε και τον πολιτικό χαρακτήρα. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας. Είναι τεχνικό το θέμα και ασφαλώς και μπορούν να βελτιωθούν οι τεχνικές λεπτομέρειες. Αλλά υπάρχουν και άλλες πολιτικές διαστάσεις. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά τη σύλληψη των πειρατών. Την δίωξή τους αντιμετωπίζουμε προβλήματα από αυτή την άποψη. Και αυτό μας εξαναγκάζει να χρησιμοποιήσουμε μέτρα αποτροπής. Και ξέρετε, αυτός ο παράγοντας της αποτροπής είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Οι επιθέσεις ε, είναι μόνο το σύμπτωμα, αν θέλετε. Η αιτία βρίσκεται κάπου αλλού. Μία πρακτική πρόταση να κάνω. Γνωρίζετε ότι οι ομάδες, ε, οι μάχες θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν και για άλλους σκοπούς πέρα από τους στρατιωτικούς. Είναι εξορισμού υποψήφοι, αν θέλετε, για τέτοια προβλήματα καταστροφών και τώρα υπάρχει και ε, μία συγκυρία περίεργη. Έχουμε τη Χιλή, την Αϊτή. Έχουμε λοιπόν τα μέσα αυτά, τα οποία όμως έχουν συλληφθεί στρατιωτικής βάσης. Αλλά πλέον έχουμε μία συγκέντρωση των πολιτικών μέσων. Πώς μπορούμε λοιπόν να δώσουμε και μια πολιτική διάσταση, διάσταση πολιτικής προστασίας σε τέτοιες ομάδες που καλούνται να επιτελέσουν ένα καθήκον όχι στρατιωτικό, ο συνδυασμό θα ήταν μια καλή ιδέα τη πολιτικής, πολιτική ε, πολιτικής της προστασίας και στρατιωτική ε, αρρωγή. Ευχαριστούμε. Θα ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Έχω ένα κατάλογο με περίπου 10 αγορητέ. Θα σα παρακαλέσω να περιοριστείτε σε ένα λεπτό περίπου, ώστε να έχουμε το χρόνο και για πυκνέ παρεμβάσει μετά. Ε, Κυρία Υπουργέ, εκ μέρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού κόμματο, σα καλωσορίζουμε εδώ και έχετε τι καλύτερε ευχέ μα για να πετύχετε τους φιλόδοξους στόχους της Ισπανικής Προεδρίας για άμυνα και ασφάλεια και για την αντίστοιχη ευρωπαϊκή πολιτική, η οποία να είναι πιο αποτελεσματική και πιο δυναμική. Χωρίς καμία επιφυλαξή συμφωνούμε με τις προσπαθίες σας κατά της πειρατείας στον Δικό όπως συζητήθηκε στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών για την επιχείρηση Αταλάντε τώρα όσον αφορά τις σχέσεις ΝΑΤΟ και, και, και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, τα συζητήσαμε με τον Γενικό Γραμματείο του ΝΑΤΟ, αλλά δεν ήρθε δυστυχώς η, η πατή εκπρόσωπος. Πέστε μας, τι πιστεύετε για τις προτάσεις που διατυπώθηκαν για διμερή σύμβαση και συμφωνία με την Τουρκία. Περισσότερη συμμετοχή στην ΚΕΠΑ της Τουρκίας και γενικότερα για χώρε που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά που συμμετέχουν σε στρατιωτικέ επιχειρήσει να είναι δυνατόν να ενταχθούν στο πλαίσιο και μηχανισμό λήψη αποφάσεων. Τι πιστεύετε για αυτή την καταρχήν συμφωνία που έγινε όσον αφορά ε, το, το, το, αεροπλανοφόρο που είπαμε και τη χρήση του αεροπλανοφόρου σε σχέση με την, με, με την οικονομική πτυχή και την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και ο κύριος Γκέιτς είπε ότι η αποστατικοποίηση δεν είναι σωστή, ότι θα πρέπει κάτι να κάνουμε και έχουμε τον αναλυστή Ρόμπιν που είπε ότι μετά τον ψυχρό πόλεμο ανέλαβε τράση η Ευρωπαϊκή Ένωση για κάποια μέτωπα που δεν ήταν πάντοτε ε, πραγματικά, δεν έκανε κάτι που ήταν ρεαλιστικό. Εσείς τι λέτε για αυτές τις δηλώσεις του Υπουργού. Ο δικαστής Βελάσκο αποφάνθηκε σε ε, καταδικαστική απόφαση ότι Έγινε συνεργασία ε, για εγκληματική δράση της ΕΤΑ με τους ΦΑΡΚ για να δολοφονήσουν στην Ισπανία τον, ε, τον, τον επικεφαλής, τον αρχηγό κράτους της Βενεζουέλας. Μας ανησυχεί η κατάσταση αυτή, αλλά και οι σχετικές δηλώσεις που ακολούθησαν. Merci, ε, Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε. Κυρία Υπουργέ, με μεγάλη ικανοποίηση διαπιστώνουμε ότι με μεγάλη προθυμία έρχεται να συζητήσουμε η Ισπανική Προεδρία. Αναφέρατε για το ρόλο της Ένωσης όσον αφορά τις κατεπίγουσες ανθρωπιστικές ε, ανάγκες όπως ε, αυτό το οποίο έγινε στην IT και όταν μόλι έγινε ο σεισμό γρήγορα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επίση είμαστε πεπισμένοι ότι θα πρέπει να βελτιωθεί ο μηχανισμό μα και έτσι να αντιδρά ακόμα καλύτερα η Ευρωπαϊκή Ένωση και να έχει καλύτερο συντονισμό. Όποτε έχουμε κάποιο είδου τόσο μεγάλε θεομηνίε προκαλούν ανθρωπιστικέ κρίσει. Μπορείτε να μα πείτε περισσότερα πράγματα πάνω στι προτάσει τη Προεδρία. Είμαι ευρωβουλευτής από την Αυστρία, αλλά στα ισπανικά θα σας πω καλώς ορίσατε. Και είστε μία από τις λίγες γυναίκες υπουργούς άμυνας στον κόσμο. Γιατί ξοχήν αντρικός τομέας είναι οι τομεί που μας απασχολούν εδώ, δηλαδή άμυνα, ασφάλεια και εξωτερικέ υποθέσει. Τρει ερωτήσει έχω κυρία Υπουργέ. Μας ε, μιλήσατε για κάτι που κατά τη γνώμη μου πρέπει να το συζητήσουμε περισσότερο, δηλαδή η πρόληψη των κρίσεων. Έχουμε επίση και τις νέες διατάξει συνθήκη τη Λισαβόνα, οι εξωτερικέ σχέσει και τα σχετικά. Για πετε μα. Πώς μπορείτε να προωθήσετε αυτές τις προτάσεις, γιατί έχουμε και άλλα ζητήματα όπως την κλιματική αλλαγή ε, και άλλα θέματα ασφάλειας που τα έχει έκθεση των ζώων που συζητούμε εδώ. Εσείς, σαν Προεδρία, τι θα κάνετε ούτως ώστε να υλοποιήσετε αυτές, ε, αυτές τις πτυχές της πολιτικής, της, δηλαδή την πρόληψη των κρίσεων, τι μπορούμε να έχουμε σαν μόνιμη δομή για αυτή τη δουλειά. Στη σελίδα 20 του κειμένου της 24 Δευτέρου. Λέτε ότι σαν Προεδρία θέλετε μια Ευρώπη πιο ισχυρή, όμως αναφέρατε εσείς ότι θα πρέπει να υπάρχει κάποια συμφωνία όλων για μια κεπά που να έχει και ένοπλες δυνάμεις. Όπω ξέρετε έχουμε έξι χώρε που είναι ουδέτερες, γι' αυτό και το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ διφορούμενο. Ε, είμαστε στην ΚΕΠΑ, αλλά είμαστε ουδέτεροι. Εσείς επομένως, ε, τι ρόλο θα μας δώσετε για εμά των, ουδετέρων χώρων. Θα έχουμε κάποιο ρόλο, εάν υπάρξει τέτοια ΚΕΠΑ με στρατό. Είπατε επίση και για τη βιομηχανία, τη σχετική με την πολιτική τη άμυνα, στρατιωτική βιομηχανία. Ο κύριο Πασχουάλ είπε ότι αυτό από πολιτική πλευρά είναι ίσω λίγο προβληματικό. Και η πρότασή σα να μειωθεί ε, να, μειωθεί ο, ο στρατός, η, η αμυντική πολιτική τέλο πάντων, να το των μελών για να συμμετέχουν περισσότερο στην ε, ευρωπαϊκή αμυντική πολιτική. Πώς θα γίνει. Τώρα, έχουμε την, ε, αυτό είπε η κυρία Άστον, έχουμε το 2006 ε, την έκθεση Μπαρνιέ για, μια, για ένα κοινό ευρωπαϊκό στρατό ή για μια δύναμη επέμβασης για ανθρωπιστικές κρίσεις. Είναι, είναι αυτό μια σωστή αφετηρία. Merci. Ευχαριστούμε. Θα έλεγα κυρία Υπουργέ να απαντήσετε σε αυτό το πρώτο γύρο ερωτήσεων για να συνεχίσουμε μετά με τους υπόλοιπους αγορητές. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Θα προσπαθήσω να σας απαντήσω μια, βέβαια δεν θα είναι πάρα πολύ εύκολο γιατί πιέζει ο χρόνο. Όσον αφορά το Συμβούλιο των Υπουργών Αμήνες. Αναφέρθηκαν κάποιοι από εσά. Υπήρξε συνένεση μετά από κάποιε και συζητήσει, είπαμε όλοι ότι είναι μια ευκαιρία τη Λισαβόνα και έτσι μπορούμε με θεσμικό τρόπο να ε, παγιώσουμε την ΚΕΠΑ. Στα πλαίσια του Συμβουλίου Εξωτερικών θα συναντιόμαστε, προβλέπει η συνθήκη. Άρα θα αποκτήσει επίσημο χαρακτήρα η συνάντησή μας και θα λαμβάνουμε κάποιες αποφάσεις που σε εθνικό επίπεδο ε, λαμβάνουν οι Υπουργοί Εθνικής Άμυνας, όπως τα της βιομηχανίας άμυνας που θέλουμε να προωθηθεί. Και ότι μόνο έτσι, αν έχουμε τέτοια ισχυρή ε, βιομηχανία άμυνας, μπορούμε να έχουμε ισχυρή πολιτική άμυνα στην Ευρώπη. Άρα θα εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία της συνήθιλης αγώνας. Επίση, θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει όσον αφορά τις στρατιωτικές ε, δυνάμεις, την πλαισιωσή του και θα πρέπει σε συνεννόηση με του Υπουργού Εξωτερικών να πρέπει να δούμε τι καινούργιε επιχειρήσει θα έχουμε, τι προλήψει κρίσεων, τι εμπλοκή, μάλλον τι συνεννόηση θα έχουμε με άλλου ε, στη διεθνή σκηνή. Και στι συναντήσει μα, επομένω, όποτε είναι δυνατόν, θα πρέπει να λαμβάνουμε κάποιε αποφάσει. Ακριβώ όπω γίνεται και σε επίπεδο εθνικό. Μια που έχουν περάσει 10 χρόνια από τότε που ξεκίνησε η ΚΕΠΑ. Νομίζω ότι τα πήγαμε καλά και εξελίσσεται αυτό το όραμα της ε, πολιτικής άμυνας και ασφάλειας για την Ένωση. Επίσης, Όσον αφορά αυτά τα οποία ρωτήσατε για την ολοκληρωμένη οπτική που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τις κρίσεις και για τις συγκρούσεις και ότι θα πρέπει Άρα, όπως έκανε και η Σουηδική, Προεδρία, θα κάνει και η Ισπανική, να προσπαθεί με στρατιωτικά και πολιτικά μέσα ολοκληρώνεται τώρα αυτό το πρόγραμμα του 2010 και θα ξεκινήσουμε ε, ένα καινούργιο πρόγραμμα ε, για 20 ετή ορίζοντα. Τώρα, όσον αφορά ε, αυτά που είπε ο κ. Αλεξάνδρ Μπέις, εμείς θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ θετικό το τι προβλέπει η συνθήκη της Λισαβόνας. Η υπηρεσία άμυνας θα είναι πάρα πολύ βασικό στοιχείο στο να εξελίξουμε την πολιτική άμυνας. Ε, επανειλημμένα έχουμε πει ότι θα πρέπει να αναπτύσσουμε τις δυνατότητές μας, να βελτιώσουμε τις επιδόσεις μας, ανάπτυξη των ε, δυνάμεων, έρευνα, προγράμματα εξοπλισμού, συνεργασία, τεχνολογία άμυνας, έρευνα του τι ισχύει στις άλλες αγορές και επομένως έτσι θεωρούμε ότι θα οριμάσει ο προβληματισμός για το τι νομικό χαρακτήρα θα έχει η υπηρεσία ασφάλειας και άμυνας. Αυτό θα ζητηθεί στο Λουξεμβούργο και θα δούμε ακριβώς πόσο μόνιμο χαρακτήρα θα έχει η, η, η, διοικητική δομή. Επίσης έχουμε κάποιες άλλες ερωτήσεις όσον αφορά την ε, επιχείρηση Αταλάντη. Ήταν η πρώτη κατά θάλασσα επιχείρηση, ε, πέτυχε ε, συνεργαστήκαμε και με το ΝΑΤΟ, με τρίτες χώρες, Κίνα και Ρωσία, συνεργασία και συντονισμός πήγε πάρα πολύ καλά. Και η επιχείρηση ήταν επιτυχής. Ε, από μόνοι μας βέβαια δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε, πρέπει να συνεργαζόμαστε και με τους άλλους, αλλά είπαμε, ήταν, πήγε, πήγε πάρα πολύ καλά. Όμως ε, δεν σταματάμε εδώ, θα πρέπει αφού περιορίσαμε την πειρατεία θα πρέπει να την ε, εκριζώσουμε τελείως στην ε, Ανατολική Αφρική. Όμως θα πρέπει να μπορούμε να δράσουμε και από ξηράς. Θα είναι επομένως στρατιωτική επιχείρηση, αλλά εμείς δεν θεωρούμε ότι η λύση είναι ε, ποτέ μόνο στρατιωτική. Επομένως, μετά από ένα χρόνο μπορούμε να βελτιώσουμε τις επιδόσεις μας στις επιχείρησεις θάλασσα στη συνεργασία με τον ΟΙΕ ορίσαμε τώρα το καινούριο επικεφαλής του επιτελείου αυτών των επιχειρήσεων και έχουμε να αντιμετωπίσουμε και τα βασικά πλοία και, και τα εξαρτώμενα από αυτά όσον αφορά τους πειρατές. Θα πρέπει να χτυπήσουμε και τα λιμάνια που πάνε και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε ε, με, με τις σχετικές χώρες για να, για να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερες δυνάμεις. Ήδη υπάρχει φρεγάτα, υπάρχουν διάφορα πολεμικά πλοία, αλλά όλο ένα και περισσότερε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση καταλαβαίνουν ότι οι καινούριε αρμοδιότητες του επικεφαλής τη επιχείρησης πρόκειται να μα βελτιώσουν τι ε, επιδόσει. Βέβαια είναι και θέμα ε, οικονομικής πλαισίωσης. Αυτό μας προσχωρεί στους ε, αρμόδιους υπουργούς. Θα πρέπει να δούμε πώς θα γίνει η χρηματοδότηση με καλύτερο τρόπο. Όμως, θα πρέπει με κάθε επιφύλαξη να δούμε τι θα κάνουμε στην ε, αποξηράς δράση. Και έτσι θα πρέπει να αποκτήσουμε τις κατάλληλες υποδομές. Αυτό προϋποθέτει δράση και συνεργασία με την Σομαλία. Αλλιώς δεν γίνεται τίποτα. Είναι πάλι πάρα πολύ σωστό για να έχει αξιοπιστία η επιχείρηση να έχουμε και την κατάλληλη νομική πλαισίωση ε, για κατασχέσεις, για φυλάκιση πειρατών, ε, ε, η δίκη τους να γίνεται όπως πρέπει, γιατί είναι κάτι το πάρα πολύ βασικό. Οπότε και αυτό και έχουμε συμφωνίες με την Κένια. Αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει μόνο η Κένια σαν, σαν χώρα με την οποία έχουμε συμφωνήσει και δεν αρκεί. Θα πρέπει να συνεχθούμε και με άλλες χώρες, θα πρέπει να δούμε πώς θα συνεννοηθούμε με Μαυρίκιο, Νοτιοαφρικανική Δημοκρατία και Τανζανία. Απευθυνθήκαμε και στο ΝΑΤΟ νομίζω ότι σε αυτή τη συγκυρία τα πάμε πάρα πολύ καλά με τον ΝΑΤΟ, ούτως ώστε να είναι δυνατόν να ε, περνάνε από δίκαιη δίκη οι συλλαμβανόμενοι πειρατές. Να υπάρχει τόσο μια κάπως μόνιμη δομή για την εκδίκαση των υποθέσεων. Επομένως, Νομίζω ότι τα πράγματα βελτιώνονται σε σχέση με το τι είχαμε στο παρελθόν. Ε, φυσικά και χρειάζεται εξυγχρονισμός των δυνάμεων που λαμβάνουν μέρος στην επιχείρηση ε, αλλά όσον αφορά πολιτικές και σταθιωτικές προσπάθειες θεωρούμε ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να προσέξει για να είναι παρούσα ε, και στις ε, έκτακτες περιπτώσεις όπως οι ανθρωπιστικές κρίσεις, όπως η ΑΕΤ. αιτήση του ΟΗΕ και της ε, αιτινής κυβέρνησης βοηθήσαμε, βοηθήσαμε με πολιτικά μέσα. Γιατρούς, υλικό, ε, με ειδικού που φρόντισαν το πώς θα υπάρχει πόσιμο νερό, ε, με διάσωση ε, ατόμων από γκρεμισμένα κτίρια. Όλα αυτά γίνανε από προσωπικό των Ισπανικών Αλλοδυναμιών. Γι' αυτό νομίζω, Πρόεδρε, ότι αυτές οι ομάδες επέμβασης είναι κάτι το οποίο έχει μεγάλη δυναμική και γι' αυτό και προσπαθούμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η χρήση αυτών των ε, ομάδων σύμφωνα με τόσα συζητήσαμε και στην ε, Μαγιόρκα. Αυτές είναι οι θέσεις της ε, Ισπανίας. Ευχαριστούμε κύριε Σαλαφράγκα για τα καλά σας λόγια και για τις ερωτήσεις σας. Το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση βεβαίως και ξέρουν ότι χρειάζεται ο κόσμος μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα είπαμε αυτά ξεκάθαρα και ευχαριστούμε που ο κύριος ε, Ρασμούσεν στην Πάλμα προσήλθε να συζητήσει και ζητήθηκε το πώς θα υπάρχει κάποια σταθεροποίηση, ε, πώς θα υπάρχει κάποια συνέχεια στα πρωτόκολλα συνεργασίας, στα επιχειρησιακά θέατρα, Υπάρχει συνεργασία και ξέρετε και στο οικοσυχοπαίδιο, Σομαλία, Αφγανιστάν ισχύει αυτό. Και ξέρουμε ότι είναι κοινή δράση και ότι έτσι πιάνουν τόπο και οι, οι οικονομικές ε, πλαισιώσεις της δράσης. Όλο ένα επομένως και επεκτείνουμε τη δράση μας και αυτό ήταν ομόφωνο. Υπάρχει η βούληση ότι μπορούμε να έχουμε ε, κοινούς ανθρώπινους πόρους με τον άτομο, κοινέ δομές και έτσι να τα πάμε καλύτερα. και με τρίτες χώρες και με διεθνείς φορείς μπορούμε να έχουμε συνεργασία και αναφέρατε το παράδειγμα της Τουρκίας είναι σημαντικός εταίρος συνεργαζόμαστε έχουμε διάφορες ε, αποστολές και επιχειρήσεις που συμμετέχουν οι Τούρκοι οπότε υπάρχει η πολιτική βούληση να συνεχιστεί αυτή η συνεργασία Ξέρετε ότι εμείς θέλουμε να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία και θα πρέπει να γίνουν σχετικέ σχετικές ε, ρυθμίσει για να συμμετάσχει στην ΚΕΠΑ. Η, η Τουρκία ήδη έχει γίνει, όπως τις περιπτώσεις που είπατε. Έτσι βλέπουμε τα πράγματα ως Προεδρία. Καλύτερη συνεργασία με διεθνείς φορείς και με άλλες χώρες. Επίσης, οι 7 χώρες, οι 27 χώρες που πήγαν στην Πάλμα, συμφωνήσανε για, για την ε, αεροπορία και θεωρήσαμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικός ο ρόλος αυτών των αποφάσεων για την βιομηχανία άμυνας Χθε, και αύριο την Παρασκευή θα συνεχιστούν οι συνεννοήσεις για κάποιους χώρους ε, για κάποιες επενδύσεις. Μιλάμε για επενδύσεις 5 δις ευρώ. υπήρξαν αυτές οι 7 χώρες που προβάλλαν κάποιο, κάποιο, κάποιο αίτημα για αυτό το, το, το αεροπλάνο που θέλουμε να κατασκευαστεί το, το μαχητικό. Ε, ήταν το κλίμα για αυτό το αίτημα. Επομένως, βοηθάμε κι εμείς, βοηθάει και η βιομηχανία, ούτως ώστε να τηρηθούν κάποια, κάποια χρονικά πλαίσια, ούτως ώστε το α400 μη να υλοποιηθεί. Ρώτησατε κάτι για τη Βενεζουέλα. Ζητήσαμε εξηγήσει όπως ξέρετε. Περιμένουμε να απαντήσει η Βενεζουέλα. Προχωρά η δικαστική έρευνα γιατί η κατάσταση είναι πάρα πολύ σοβαρή και συμφωνώ σε όσα είπατε ο κύριος Γκέιτς. Ξέρει για τις υποσχέσεις, τις δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για κάποιες συνεργασίες, κυρίως όσον αφορά τα θέατρα επιχειρήσεων. Τα πράγματα είναι πιο δύσκολα από ό,τι τουλάχιστον τελευταία 20 ετία. Ε, αυτό ισχύει για το Αφγανιστάν, το δε 40% των νέων ενόπλων δυνάμεων προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οπότε ξέρουν. Ξέρει τι προσπάθεια καταβάλουμε εμείς στο Αφγανιστάν. Για την Ιουσαφ θέλουμε να υπάρχει σταθερότητα και ανασυγκρότηση. και όλοι τι Ευρωπαϊκή Ένωση που, είμαστε, που εκπροσωπούμαστε στο ΝΑΤΟ προσπαθούμε να χαράξουμε τη νέα στρατηγική. Νέα στρατηγική. Νέα στρατηγική που ξεκίνησε από τότε που ανέλαβε η κυβέρνηση Ομπάμα. Θέλουμε επομένω να πάρουν στα χέρια του τι διάφορε δομέ εκεί η Αφγανία. Αφγανοποίηση το λέμε και θεωρούμε ότι σύντομα θα υλοποιηθούν οι ιδέες μας. Όμως παραλαμβάνω, είναι η πιο σκληρή, η πιο δύσκολη αποστολή που έχουμε αναλάβει. Κύριε Νόνια. Α, Λούντσικ. Ναι. Σας ευχαριστούμε. Ήταν πολύ σωστή αυτή η ερώτηση που κάνατε που αφορά την πρόληψη των κρίσεων. Για μας είναι προτεραιότητα όπως και η Αταλάντη. Η απάντηση έγκυται σε μια ολοκληρωμένη πολιτική. Προσπάθειες διπλωματικές, οικονομικές, αναπτυξιακές και στρατιωτικές. Α, όταν χρειάζεται. Άρα χρειάζεται μια στιβαρή εξωτερική πολιτική από την Ένωση που δεν μπορεί παρά να στηρίζεται σε ένα τέτοιο ολοκληρωμένο όραμα και άποψη των πραγμάτων. Η δε συνήκη της Λισαβόνας μας δίνει τη δυνατότητα, γι' αυτό και προβλέπει την ύπατη εκπρόσωπο. Και έτσι να υπάρχει τέτοιου είδους αντιμετώπιση μέσω της Κομισιόν για την πολιτική αυτή. ένα πρόσωπο είναι και μπορεί όμως όλα αυτά να τα όλες αυτές τις διαφορετικές πτυχές που χρειάζονται να τις αναλάβει. Άρα έχουμε κοινή εκπρόσωπο, κοινή άποψη επομένω και για την πρόληψη των κρίσεων. Τώρα όσον αφορά την ε, πάγια, διαρθρωμένη, δομημένη συνεργασία. Είμαστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί όσον αφορά την υπόθεση αυτή. Αλλά όσο πιο νωρίς προχωρήσουμε τόσο το καλύτερο. Να μας βοηθήσει το Κοινοβούλιο στο πώς θα σχεδιαστεί αυτή η δομημένη συνεργασία. Θέλουμε όμως να είμαστε επιφυλακτικοί γιατί πάντοτε είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει συνένεση. Δεν θέλουμε να υπάρχουν δύο ταχύτητες και κάποιο να περιθωριοποιείται, κάποιο να μην συμμετέχει. Να συμμετέχουν βέβαια όλοι όσοι θέλουν έτσι την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή συζητούμε και αυτή προσπαθούμε με προσοχή να προωθήσουμε αυτή τη συνεργασία. Οι 27 θέλουμε να υπάρξει μια τέτοια συνεργασία. με την υπατή εκπρόσωπο συνεργαζόμαστε σαν Προεδρία. Ευθύνη μας είναι να βοηθήσουμε να υλοποιηθούν αυτά που προβλέπει η Συνθήκη της Λισαβόνας για την ε, Ευρωπαϊκή Αμυντική Πολιτική. Γι' αυτό και κάναμε το σεμινάριο. Ούτως ώστε τα υπέρ και τα κατά ειδικοί να μας τα εξηγήσουν και να δούμε πώς θα γίνει αυτή η δομημένη συνεργασία. Νομίζω ότι απάντησα στα περισσότερα που ρωτήσατε. Ό,τι άλλο θέλετε, στη διάθεσή σα. Ευχαριστούμε κυρία Υπουργέ, απαντήσατε τόσο διεξοδικά. Αυτό σημαίνει όμω για όλου του υπόλοιπου συναδέλφου που έχουν ζητήσει το λόγο θα πρέπει να περιοριστείτε ιδιαίτερω. Θα πρέπει να είστε συντομότατοι. Καλή επιτυχία για το επόμενο δίμηνο που σας απομένει, όσους, μην, γιατί το διάστημα που θα έχετε την Προεδρία είναι πάρα πολύ σημαντικό στον αφορά τον έλεγχο τη διάδοση των πυρηνικών. Το Μάιο νομίζω θα αναφερθεί η σχετική συνθήκη τη μη διάδοση των πυρηνικών και ταυτόχρονα θα πρέπει να δούμε το πόσο όλοι ανησυχούμε όσον αφορά τα πυρηνικά του Ιράν. Ήδη έχουν κυκλοφορήσει σχέδια κειμένων του Συμβούλιο Ασφάλειας για κυρώσεις κατά του Ιράν. Αναφέρατε το Αφγανιστάν και τις ε, εκεί ευρωπαϊκές δυνάμεις που είναι ως δυνάμεις κατών μελών και όχι ως δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμφωνώ μαζί σας. Είναι σημαντικό να μας βοηθά το Πακιστάν. Εκεί ε, καταφεύγουν οι Ταλιμπάν, ε, στο Βαζιριστάν, βορρά, νότο, τον Ιούνιο. Θα γίνει συνάντηση ε, και με την Τσεχική Προεδρία, όπου θα συναντηθούμε με τους Πακιστανούς ίσως αργότερα συνεργαστεί και η Ισπανική Προεδρία. Είναι πάρα πολύ σημαντική συνεργασία με το Πακιστάν. Γιατί και το Παγιστάν έχει πυρηνικά όπλα. Ευχαριστούμε κύριος Γιάννης. Ε, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Πρώτα-πρώτα, συγχαρητήρια κυρία Υπουργέ για δύο λόγους. Πάρα πολύ πλήρη είναι τα όσα μας είπατε και θέλω τώρα να ζητήσω να μου διευκρινίσετε κάποια ζητήματα. Το α200 μη, το, την Αταλάντη, αλλά σήμερα οι Ισπανικές Προεδρίες λένε ότι στον Ταβός είπατε ότι μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο. Δεν μας εκπλήσει αυτό. Γιατί θα εκπλήσει κάποιους άλλους που ξέρουν λιγότερο τη χώρα μας. Αλλά θεωρούμε ότι όντως μπορούμε να βοηθήσουμε στο να αλλάξει ο κόσμος. Τώρα, συγκεκριμένη ερώτηση. Εδώ στην Υποπιτροπή Άμυνας θεωρούμε ότι η ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή πολιτική άμυνας και ασφάλειας θα πρέπει να προβάλλεται προς τον υπόλοιπο κόσμο ως μια πολιτική αποτρεπτική και αξιόπιστη. Οι άλλοι μας κρίνουν, δεν κρίνουμε εμείς τον εαυτό μας. Αν επομένως οι άλλοι θεωρούν ότι βοηθάμε στη τήρηση ειρήνη, έχουμε αποτρεπτικό ρόλο. Ε, έτσι θα μας παίρνουν στα σοβαρά. Τότε επομένω να θεωρήσουμε ότι υπάρχει πολιτική ασφάλειας και άμυνας που αξίζει. Ε, δεν τα είχαμε πάει καλά στην αρχή, όσον αφορά την πολιτική, είχαμε το φιάσκο στην ε, Γαλλική Εθνική Συνέλευση. Και όμως τα τελευταία δέκα χρόνια και με τη βοήθεια του Σολάνα σιγά σιγά την οικοδομούμε αυτή την πολιτική σαν μια γενική ομπρέλα. Έχουμε βέβαια την συνθήκη της Λισαβόνας που προσδίδει και στο Ευρωκοινοβούλιο κάποιες αρμοδιότητες. Όλοι οι Υπουργοί Άμυνας των κρατών μελών είπαμε ότι συμφωνούν. Όμως, ξέρουμε ότι κάποια κρατημέλη και παλιά και καινούργια που δεν συμφωνούν όσον αφορά την αντίληψη της ασφάλειας και άμυνας που μας εκθέσατε, δηλαδή το να κοινοτικοποιηθεί η ΚΕΠΑ. Και επομένως υπάρχει εδώ ένας φραγμός στην επιθυμητή εξέλιξη. Οι συνάδελφοί σας, οι ομόλογοί σας, δεν συμφωνούν όλοι. Ευχαριστούμε κύριο Ζωμέβα. Ευχαριστώ και εγώ να σας ε, συγχαρώ και έχω δύο ερωτήσει, μια που πιέζει ο χρόνος, πρώτα-πρώτα, για την διάδοση των πυρηνικών και σε σχέση με τα συμβατικά όπλα, είπαμε ότι προσπαθούμε να ρυθμίσουμε τα του εμπορίου των όπλων. Εσείς τι θέση παίρνετε. Τι θέση παίρνει η Ευρώπη. Άλλη ερώτηση. Έχουμε τώρα την δέκατη επέτειο του ψηφίσμου 13-25 του ΟΗΕ όσον αφορά το ρόλο της γυναίκας στους πολέμους. Και το 2008 είχαμε κι άλλο ένα ψήφισμα όσον αφορά τη χρήση του βιασμού ως όπλο. Ξέρω ότι η Ισπανία έχει ασχοληθεί ως Προεδρία, αλλά πέστε μας, τι θα κάνετε συγκεκριμένα ούτως ώστε να υλοποιήσετε αυτά τα δύο ψηφίσματα. Ευχαριστούμε κύριο Σκέλαμ. Ευχαριστώ. Κυρία Υπουργέ, σας ευχαριστούμε που επιβεβαιώσατε τον σημαντικό ρόλο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφαλείας. Άμυνας μάλλον, συγγνώμη. Αυτή ήταν και η δική μου ερώτηση, γιατί μέχρι τώρα τα στοιχεία που μας δώσατε ήταν ε, θετικά. Και σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της συνθήκης της Λισαβόνας, νομίζω ένα σημαντικό σκέλος είναι ο συντονισμός. Και θέλω να ρωτήσω ακριβώς πώς σκοπεύετε να συντονιστείτε σε εβδομαδιαίο επίπεδο, σε εβδομαδιαία βάση, σε συνεργασία με την πρόσωπο και με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους δικούς τους ε, ηθήνοντες. Και ήθελα και την άποψή σας για ένα άλλο θέμα. Για την πώληση τεχνολογικών μέσων εχμής σε τρίτα μέρη. Είναι αυτό μέρος ή θα έπρεπε να είναι μέρος της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το να απολυθούν ας πούμε ελικόπτερα προς την Ρωσία, μια χώρα που είναι απειλητική προς τις γειτόνες της ιδίως τον τελευταίο καιρό δεν έχει σεβαστεί τις ρήτρες όλων των συμφωνιών της και το περασμένο φθινόπωρο έφερε εις πέρας και στρατιωτικές ασκήσεις και κάποιες φορές απειλώντας και κάτι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι τέτοιο λοιπόν δεν θα έπρεπε να το δούμε καλύτερα στα πλαίσια των κοινών μας πολιτικών. Ευχαριστούμε κυρία Γκόμες. Καλώς ορίσατε κυρία. Και εγώ, όπως και εσείς, είμαστε γυναίκες που ασχολιόμαστε με αυτή την πολιτική να έχουν περισσότερη ασφάλεια και ειρήνη στον κόσμο. στο, στο πλαίσιο αυτών, επομένως, των σχέσεων ΝΑΤΟ-ΕΕ και εν ώψη της συνάντησης του Νοεμβρίου της Λισαβόνας με τον ΝΑΤΟ προσπαθούμε να έχουμε μια ευρωπαϊκή θέση. Να μην λέει ο καθένας το δικό του. Να βγούμαστε με μία φωνή. Έχουμε τα όπλα μαζικής καταστροφής. Μεγάλη απειλή. Η κυβέρνηση Ομπάμα έλαβε κάποιες ε, αποφάσεις αλλαγής πολιτικής και έχουμε εδώ πέρα τώρα και το θέμα των πυρηνικών όπλων και όπως είπε και κάποιος άλλος συνάδελφος η Ισπανική Προεδρία έχει κάνει πάρα πολλά όσον αφορά το, τα ψηφίσματα του ΟΗΕ και είναι πάρα πολύ σημαντικό να δουλέψουμε ούτως ώστε να δούμε τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το Κονγκό, που είναι μια χώρα όπου έχουμε πάρα πολλές αποστολές, άρτεμις κλπ. Έχουμε πολλά προβλήματα ε, όπου χρησιμοποιεί το βιασμό ως όπλο και θα πρέπει να δούμε πώς θα είμαστε πιο αποτελεσματικοί που δεν είμαστε. Τέλος για τη Σομαλία. Σωστά είπατε ότι, ότι από ξηρά το πρόβλημα. Μιλήσατε για τις προσπάθειες της κατάρτισης των δυνάμεων εκεί. Ξέρουμε όμως όλοι ότι στη Σομαλία δεν υπάρχει κράτος. υπάρχει μια κυβέρνηση σε εμβριώδη κατάσταση Πώς θα γίνει η κατάρτιση των νόπλων δυνάμεων. Πρέπει να προηγηθεί ενίσχυση των κρατικών δομών. Μην μές πως μας στο κενό. γιατί είναι δύσκολο θέμα, είναι πολυδάπανο. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να προσπαθήσουμε εκεί, γιατί η χώρα αυτή στην πρώτη γραμμή της, της αντιμετώπισης της τρομοκρατίας. Κύριε Υπουργέ. Por ejemplo, por, por, por esta última, mire, una, uno de nuestros mayores riesgos ahora mismo son los estados fallidos. Y Όντως, εκεί που δεν υπάρχει κράτος, ε, υπάρχει πρόβλημα και ε, κάθε φορά, κάθε, κάθε μέρα το, το, το, το, βλέπουμε και το διαπιστώνουμε αυτό. Και ξέρουμε ότι και η κατά ξηράν επιχείρηση είναι πάρα πολύ βασικό. Το ξέρουμε και εμείς, το, το ξέρουν και οι υπόλοιποι διεθνείς παράγοντες. και θα πρέπει να δούμε πώς παρά την μεταβατική κατάσταση στην Σομαλία θα γίνει αυτή η εκπαίδευση των ενόπλων δυνάμεων. Πρέπει να υπάρχει ένα, ένα, ένα μήνυμο υποδομών και ασφάλειας για να δουλέψουμε. Άρα, ο επικεφαλής του επιτελείου, ο επικεφαλής της ε, στρατιωτικής εκπαίδευσης συνεργάζονται με την ε, μεταβατική ε, κυβέρνηση της χώρας. Ξέρουν πόσο σημαντικό είναι, πόσο σημαντικό είναι για την παγκόσμια ασφάλεια. Και αυτό αφορά κάθε πεδίο σύγκρουσης, όπως και το Αφγανιστάν τότε στο Αφγανιστάν, παλιότερα τώρα στην ε, Σομαλία. Οι έλεγχοι που γίνονται. Οπότε χρειάζεται ένας μηχανισμός επιλογής, ε, στρατολόγησης, η αμοιβέ, η χρηματοδότηση. Όλα αυτά τα έχουμε δει και αλλού. Και ευθύ εξ αρχή ήταν σαφέ ότι και στη Σομαλία έτσι θα γίνουν τα πράγματα. Ο Διεθνή Οργανισμό Ατομική Ενέργεια φυσικά και ανησυχεί για την κατάσταση στο Ιράν. Και εμεί βέβαια θέλουμε πρώτα-πρώτα να υπάρχει διάλογο, αλλά δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τις κυρώσεις εάν δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις της η χώρα αυτή. Χρειάζονται μέτρα. Και βέβαια το Συμβούλιο Ασφαλείας θα αποφασίσει για το τι μέτρα θα ληφθούν. Δεν μπορούμε παρά να συμφωνήσουμε με τον Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας. Επίσης, όσον αφορά την αναδιορίση της συνθήκης για τη Μηδιάδοση των πυρηνικών, προσπαθούμε να συμφωνήσουμε επίση με την πολιτική χρήση της ατομικής ενέργειας, ε, με την μη διάδοση των πυρνικών, ε, με τη συνάντηση κορυφής τώρα για το Πακιστάν. Ε, ήταν μια άλλη ερώτηση, όπως σωστά το είπατε, θα είναι η δεύτερη συνάντηση ε, γιατί προηγήθηκε και επί Σουηδικής Προεδρίας μια συνάντηση κορυφής. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η περιοχή, είναι πάρα πολύ σημαντική η συνεννόησή μας για τη σταθερότητα στην περιοχή εκείνη. Θα πρέπει να είμαστε συνεπεί στην πολιτική μας, την αντιτρομοκρατική, θα πρέπει να είμαστε συνεπεί και στην οικονομική συνεργασία ε, και στα θέματα παιδείας. Ε, εκεί κατευθύνεται η αρρωγή μας προς τη χώρα αυτή. και... και... Είναι μια διαδικασία που συνεχίζεται, δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι τέλειωσε εδώ αυτή η εξέλιξη. Με, για, τη χώρα αυτή τώρα μας είπατε κύριε Γκόμες για την χρήση του βιασμού ως, όπλου σε έναν πόλεμο όλη η διαδρομή της κυβέρνησης Σταπατέρο ε, ήταν, είχε ως προτεραιότητα την προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών και γι' αυτό θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το να προστατεύσουμε γυναίκες και ανηλίκους που υφίστανται και οι και η δε την βία ίστις τις ε, τις τις ε, συγκρούσεις και προσπαθούμε να ελοπίσουμε το 1325 το ψήφισμα και προσπαθούμε επίσης ε, την προσπάθειά μας αυτή να τη συμμερίζονται και άλλες στη διεθνή σκηνή. Επίσης, κυρία Γκόμες, κάτι είπατε για το Κόγκο. Έχουμε δύο αποστολές στο Κόγκο ε, σε σχέση με την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταβάλλεται προσπάθεια εκεί πέρα. Ε, συνολικά είχαμε τέσσερις όπως που έχουμε κάνει. Συνεργαζόμαστε με την αστυνομία εκεί, με, τις, με τον ΟΗΕ, πώς να αντιμετωπίσουμε τους βιασμούς που είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Και ξέρουμε ότι στη σημερινή συγκυρία θα πρέπει να δούμε τι γίνεται όσον αφορά τη σταθεροποίηση της κατάστασης στη χώρα. Γιατί γνωρίζουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει συνειδητοποίηση του τι γίνεται εκεί από, από τον πόλεμο, από την, ε, τη δυστυχία που χτυπήσει τον κόσμο. Προσπαθούμε επομένω και με πολιτικά και στρατιωτικά μέσα κάτι να κάνουμε. Θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προσπαθήσει και η Ισπανία επομένως συνεχίζει ευρωπαϊκές προσπάθειες για το Κονγκό. Θέλουμε επομένως να υπάρχει έγκαιρη προειδοποίηση, να υπάρχει πρόληψη για τις κρίσεις. Ελπίζουμε να τα καταφέρουμε. Ελπίζω, Πρόεδρε, ότι απάντησα. Α, Κύριε Γιάννη, σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Ο καθένας κάνει ό,τι μπορεί. Και... Νομίζω ότι 27 συμφωνήσαμε. Εντάξει, ο καθένας ε, όποτε μπορεί μιλάει φορτισμένο συστηματικά ή μη φορτισμένος, πάντως όλοι θέλουμε ισχυρή Ευρώπη. Στο πλάι του ΟΗΕ και των άλλων διεθνών οργανισμών. Συνεργασία. Είναι θέματα που μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Βρισκόμαστε σε φάση μεταβατική, όσον αφορά και τον ΝΑΤΟ και τον εαυτό μας για το πώς βλέπουμε τα πράγματα. Αλλά θέλουμε ότι είμαστε της Λισαβόνας θα είμαστε ενισχυμένοι με καλύτερη συνεργασία και πέρα από τις ε, δηλώσεις του καθενός, οι 27 συμφωνούμε. Και σε σχέση με το ΝΑΤΟ. Όχι, όχι, υπήρξε σχεδόν ομοφωνία. Πολιτική βούληση να προχωρήσουμε ενωμένοι. Να έχουν θεσμικό χαρακτήρα αυτές οι συναντήσεις των ε, Υπουργών Άμυνας. Και ό,τι συμφωνούμε να είναι απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και έτσι να είναι προβλήμα μα έξω το όραμά μας για ασφάλεια και ειρήνη. Κυρία Υπουργέ, σας ευχαριστούμε. Ξέρω ότι <clears throat> έχουμε ξεπεράσει λίγο το κανονικό μας ωράριο, αλλά θα μπορούσατε να απαντήσετε σε λίγες ακόμα ερωτήσεις για να μην μείνει κανείς ε, με την ερώτηση του αναπάντητη. Ο κύριος Λίζα. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσω για τις πολύ συγκεκριμένες απαντήσεις που μας δώσατε και για τις προτεραιότητες που έχετε θέσει, πολύ σημαντικές. Συχνά ακούμε πάρα πολλούς να μιλούν για δεκάδες ε, προτεραιότητες, το οποίο σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικά προτεραιότητες. Μου αρέσει λοιπόν το γεγονός ότι εσείς αναφέρατε κάποιες περιορισμένες και συγκεκριμένες ε, προτεραιότητες για την υποεπιτροπή μας. Η συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ είναι ουσιώδης σε ό,τι αφορά θέματα ασφάλειας. Αλλά, Υπουργέ, να σας ρωτήσω, θεωρείτε ότι η συνεργασία αυτή μεταξύ ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να λάβει νέο θεσμικό πλαίσιο. Ο Πολωνός υπουργό Άμυνας, ο κ. Πλέχτη, μίλησε για ενδεχόμενη ε, τροποποίηση της Συμφωνίας του Βερολίνου. Επίσης, είπατε ότι η Βοσνία και η αναφερθήκατε μάλλον στη Βοσνία και Ζεγοβίνη, θεωρείτε ότι θα πρέπει να οριστεί μια συγκεκριμένη ημερομηνία για την ε, αποστολή. κύριος Μενέντες. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλημέρα, κυρία Υπουργέ. Εδώ, εδώ είμαι. Εδώ είμαι, στα δεξιά σας. Εδώ, εδώ. Ναι, παίρνω και εγώ το λόγο. Πάντω, εσεί στην αρχή, κάποια στιγμή στη στάση μα είπατε, είπατε για του ε, ιδρυτέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί είχαμε και κάποιον άλλο όμω ε, φημισμένο. Ήταν ο Όλοφ Πάλμιο, τότε πρωθυπουργό τη Σουηδία, που έλεγε ότι η καλύτερη πολιτική τη Άμυνα είναι μία εύστοχη πολιτική εξωτερική. Πάρα πολύ σωστά επίση για την πειρατεία είπατε ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό το πρόβλημα κατά θάλασσα. Ο, και εγώ όμω η λύση βρίσκεται στην ξηρά. Θεωρώ ότι. Είναι και πολιτικό το πρόβλημα. Είναι θέμα ασφάλεια, ε, αλλά καταρχήν είναι πολιτικό το θέμα της ε, πειρατείας. Γιατί ε, πρόβλημα είναι για τη λύση του προβλήματος, φραγμός λύση του προβλήματος είναι αυτό που είπαμε ότι δεν υπάρχει κάτω στη Σομαλία. Δεν θα πρέπει να έχουμε μια δόκιμη, ολοκληρωμένη, ε, πλήρη συνεργασία. Για εξωτερικά για άμυνα και έτσι να κάνουμε πραγματικότητα αυτές τις ρίσεις του Όλαφ Πάλμα. Θα ξεκινήσω από την τελευταία ερώτηση. Α, όχι, συμπαθάτε με, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε, κύριο Λουάν, για να κλείσουμε. Ευχαριστώ και εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω Υπουργέ για την ε, πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση και τα πολύ ενδιαφέροντα σχόλια που κάνατε. Αναφερθήκατε σε πολλά μέτρα πρόληψης. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί η πρόληψη ασφαλώς είναι πιο αποτελεσματική από την εκ των υστέρων ε, παρέμβαση. Αναφορικά με την αποδοτικότητα της ανάπτυξης των στρατιωτικών δυνάμεων. Ωστόσο, η αποτελεσματικότητα των δυνάμεων αυτών γιατί μεταξύ της στιγμής που ξεσπάει μια κρίση και της παρέμβαση μιας ε, δύναμη, συνήθω συνήθως τρει τέσσερι μήνες. Ίσως θα μπορούσατε να αναφερθείτε και να συζητήσετε έναν τρόπο κατά τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να αναπτύξει ένοπλε ένοπλες δυνάμεις ανεξάρτητα από το που εκπαιδεύονται. Να υπάρχει δηλαδή έτοιμος ένας μικρός στρατός αν θέλετε, ο οποίος θα είναι σε θέση να παρέμβει άμεσα. Ίσως το θέμα αυτό είναι πολιτικό ευαίσθητο σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά δεν θεωρείτε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ θα πρέπει να εξετάσουν την εφικτότητα της λύσης αυτής. Και κατά δεύτερον θα ήθελα να τονίσω ότι το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι σχετικοί θεσμοί φαίνεται να αλληλεπικαλύπτονται στα καθήκοντά τους θα μπορούσαμε να διαμορφώσουμε με πιο αποδοτικό τρόπο τη συνεργασία μεταξύ Ένωση και ΝΑΤΟ. Όπω είπα, θα αρχίσω με την τελευταία ερώτηση, την πρώτη τελευταία τέλο πάντων. Δέκα μέρε θέλουμε να έχουμε την ανάπτυξη των δυνάμεων ταχεία, των ομάδων ταχεία επέμβαση, ούτω ώστε να είναι ένα πραγματικό εργαλείο Πολλέ φορέ όμω είναι τέτοια θεομηνία που οι δέκα μέρες ε, είναι πάρα πολύ αργά. Ε, Εμεί α πούμε θέλουμε να έχουμε για την ΑΕΤ ήταν άμεση η, η αποστολή γιατί έπρεπε να πάνε στα ερήπια, να μεταφέρουν τα πτώματα κλπ. Και το θέμα είναι τι θα γίνει με αυτέ τι ομάδε. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε αυτό το δεκαήμερο γιατί για να έχουμε αποτελεσματικότητα θα πρέπει να ενεργούσαμε πολύ πιο γρήγορα. Ακριβώς έτσι το είδε το θέμα η Ισπανική Προεδρία. Έχει το NRF, του ΝΑΤΟ, αντίστοιχα για τις θεομηνίε, για τα groups αυτά. Το θέμα είναι όμως κατά πόσο ε, αυτές οι ομάδες μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε άλλες περιπτώσεις. Επίσης μιλήσαμε για το ότι θα πρέπει να έχουμε βελτίωση και αναβάθμιση των σχέσεων με το ΝΑΤΟ. Και κατά πόσο θα υπάρχει αντιστοίχηση κάθε φορά ε, πολιτικής με στρατιωτική παρουσία του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. γι' αυτό σου ήταν πάρα πολύ δημιουργική και ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ίσως ε, από τις πιο σοβαρές, πιο πλούσιες συζητήσεις που έχω δει σε τέτοιο επίπεδο. Και κατέβασαν στο τραπέζι οι Υπουργοί όλα αυτά τα θέματα για να μπορέσουμε να δούμε τι θα κάνουμε. Κάποιο είπε για το Βερολίνο ΣΥΝ, ναι αυτό ισχύει, αλλά θα πρέπει να υπάρχει ένα σταθερό πλαίσιο Α, έφυγε ο κύριος ε, που το ρώτησε. Και επομένω υπάρχει αυτό το πλαίσιο ότι θα ρυθμίζει τις σχέσεις των δύο φορέων όταν ε, και οι δύο κάπου επεμβαίνουν. Θα πρέπει να γίνει συζήτηση, θα πρέπει να προβληματιστούμε και να υπάρξει κάποιο πρωτόκολλο συνεργασίας. Καλύτερο. γιατί έχουμε διάφορους συνδυασμούς ε, στρατιωτική δράση και των δύο ή του ενός μόνο ή πολιτική δράση και όλα αυτά να κρίνονται από τους Υπουργούς Άμυνας της Ένωσης. Βοσνία Ριτσεχοβίνη. Θα κρυθεί και θα κανονιστεί το τι θα γίνει στο Λουξεμβούργο. γιατί ακριβώ είναι εύστοχο, για να, για, να, για να είναι εύστοχη μια αποστολή θα πρέπει να είναι εύστοχη η έναρξη αλλά και η λήξη της. Αυτό θα κρυφθεί στο Λουξεμβούργο. Η στατιωτική επιχείρηση επί τη βάση του Ντέιτον έκλεισε τον κύκλο τη. Άρα θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει και να κάνουμε αυτό που τελικά ζητούν οι αρχέ τη χώρα. Βοήθεια για το Υπουργείο Άμυνα και βοήθεια στη δημιουργία ενοπλών δυνάμεων. Στο Λουξεμβούργο μπορώ να σας πω ότι έχουμε, ε, όπως είπαμε στη Μαγιόρκα, θα συνοηθούμε την Κομισιόν και θα ολοκληρώσουμε την στρατιωτική επιχείρηση. Αυτό ζητάνε. Ε, είναι και το θέμα των εκλογών στη Βοσνία. Και έτσι θα συνεχιστεί η διαδρομή, σύμφωνα με τα λόγια του Πάλμα. Επίσης είπαμε και για την καταθάλασσα επιχείρηση στην Σομαλία. Και εκεί δράσαμε πάρα πολύ σωστά γιατί μπορούσαμε να αποσπάσουμε από τον ΟΗΕ τα ψηφίσματα που χρειαζόντουσαν για την επιχείρηση. Ξέρετε, αυτές οι κυκλικά αναλασσόμενε προεδρίες δεν έχουν τόσο χρόνο χρειάζεται βέβαια. Η συνήθεια Λισαβόνα βοηθάει. όσον αφορά την αποτρεπτική πολιτική μας. Γιατί έχουμε την είπατε εκπρόσωπο. έχουμε σαν Υπουργείο Εξωτερικών και σαν Υπουργείο Άμυνα. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ για αυτή την ιδιαίτερα διεξοδική παρουσίαση, για την προθυμία σας να απαντήσετε σε όλους. Θα έχουμε και άλλες ευκαιρίες να σας ξαναδούμε κατά τη διάρκεια αυτού του εξαμήνου και προς το τέλος της Ισπανικής Προεδρίας ούτως ή άλλως. Είστε πάντοτε καλοδεχούμενοι εδώ. Σας ευχαριστούμε λοιπόν. Πιστεύω ότι δώσατε απαντήσεις σε όλα πραγματικά τα ερωτήματα που τέθηκαν. Σας ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ και να ευχαριστήσω τον συνάδελφο για την έκθεσή του για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Άμυνας. Ανυπομονώ να δω και το ε, κείμενο που θα συνταχθεί. Σας ευχαριστώ για σας ό,τι κάνετε και γιατί θα είμαστε κοντά σας στην Ισπανική Προεδρία. Ευχαριστώ.